Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το σχέδιο έκθεσης που τροποποιεί τον κανονισμό 1303 του 2013 όσον αφορά ορισμένε διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρέ δυσκολίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Το σχέδιο έκθεσης που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά το άρθρο 24 και το άρθρο 123 του ε, Κανονισμού Περικοινών Διατάξεων για υψηλότερα ποσοστά σύγχρηματοδότηση σε χώρες που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί ε, το χρονικό διάστημα. Η πρόταση αυτή δεν αναμένεται να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις και το άρθρο 24 του Κανονισμού Περί Διατάξεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις πληρωμές, να κάνει top-ups σε κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ε, βρίσκονται υπό ε, οικονομική ε, βοήθεια. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που λαμβάνει αυξημένη συγχρηματοδότηση μέχρι το τέλος του Ιουνίου φέτος. Το άρθρο προβλέπει υψηλότερε πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει να συνεχίσουν οι αυξημένε πληρωμές σε οποιοδήποτε κράτο μέλος ε, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας που απολαμβάνει οικονομικής ε, σύνδρομη μετά τις 30 Ιουνίου 2016 για την περίοδο που βρίσκεται υπό το μηχανισμό στήριξη χωρί να γίνουν τροποποίησεις ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Λάβαμε την πρόταση πριν την τελευταία μας συνεδρίαση τον Ιούλιο. Είμαι προσωπικά εισηγήτρια <coughs> για την Επιτροπή μας. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες επιτροπές, μόνο η Επιτροπή Αλληλείας και η ΕΚΟΝ ε, εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολή γνωμοδότησης, όμως δεν θα υποβάλουν, θα καταρτήσουν μάλλον γνωμοδότηση, αλλά θα στείλουν επιστολή. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, μάλλον θα, θα αποστείλει μια επιστολή. Οι υπόλοιπε επιτροπές, ε, Τραν, Κάλτα, Γκριφέμ και Ήτρε, ανέφεραν ότι δεν θα καταρτήσουν γνωμοδοτήσεις, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν έχει αποφασίσει τη θέση της μέχρι τώρα. Έτσι έχουν τα πράγματα με τις άλλες επιτροπές. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσης που προετοίμασα. Σκοπός λοιπόν της νομοθετικής πρότασης είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από τη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση να συνεχίσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί η αυξημένη συγχρηματοδότηση στα ποσοστά του 85% για την Κύπρο, να παραταθεί ο μηχανισμός top-up που ε, για την Ελλάδα και το άρθρο 4 του, 24 ε, του κοινωνισμού, ε, Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων προβλέπει ότι το κράτος μέλος το οποίο έχει προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες και οι χώρες οι οποίες έχουν λάβει στο παρελθόν ε, οικονομική στήριξη και βρίσκονται σε προγράμματα προσαρμογή από το 2013 και έπειτα ε, θα έχουν αυξημένες πληρωμές κατά 10%, το λεγόμενο top-up. Μετά, από, ε, αυτές οι πληρωμές θα προκύψουν από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Θάλασσας και Αλίας, Ανάπτυξη Τεπέθρου, και το ESF. Μέχρι το 2016 η Διελλάδα ήταν η μόνη χώρα υπό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Το άρθρο 120 του κανονισμού προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα σε κάθε ένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που ε, στηρίζονται από το ESF και το ERTF στην Κύπρο θα ε, ανέρχεται στο 85% αντί για 50% που ε, ισχύει για τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Ο κανονισμός προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτούς τους δύο κανονισμούς και εάν χρειάζεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 έτσι ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράταση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση. Η Κύπρος παρέτεινε το πρόγραμμα προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016, ωστόσο για να Βγήκε. Ωστόσο, δεδομένης της ε, πρόσθετης όθησης που χρειάζεται για να ανακάμψει η οικονομία της, Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 85% για την Κύπρο μέχρι τα τέλη του ε, πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Αυτό θα ε, ελαφρύνει τον προπολογισμό της Κύπρου κατά 99 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την παράταση του μηχανισμού top-up αναμένεται αύξηση πληρωμών κατά 10% μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και αυτό το top-up θα οδηγήσει σε ελάφρυνση δημοσιονομικών πιέσεων και θα παρέχει μεγαλύτερη ρευστότητα στις ε, άμεσες επενδύσεις. Μέχρι το 2015, εξαιτίας αυτών των διατάξεων, η Ελλάδα έλαβε 1,3 δις νωρίτερα από ό,τι ε, βλεπόταν. Αυτό επιτρέπει τα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα να μπορέσουν να ε, δρομολογηθούν συντομότερα έτσι ώστε να ε, είναι προς όφελος της ε, ελληνικής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει λοιπόν παράταση του μηχανισμού ΤΟΠΑ πέρα από τον Ιούνιο του 2006 έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να ε, ορθοποδήσει και να ε, μπει στο δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη. Στα πλαίσια λοιπόν της ιδιαίτερας μου συζητήτριας για το θέμα αυτό, προτείνω η πρόταση της Κομισιόν να εγκριθεί ως θέση του Κοινοβουλίου χωρίς τροποποίησεις. Σας προτείνω επίσης η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παραπέμψει το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο ξανά εφόσον σκοπεύει να τροποποιήσει σημαντικά την πρόταση ή να την αντικαταστήσει με κάποιο άλλο κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο έκθεσης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Δεν τους βλέπω όμως στην αίθουσα. Η κυρία Βέστφαλ. Η κυρία Βέστφαλ θα μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Κρέλ. Να σας πω ότι η κυρία Κρέλ απουσιάζει αυτή τη στιγμή από την αίθουσα. Μου έστειλε όμως ένα μήνυμα ενημερώνοντά με ότι ως σκιώδης εισηγήτρια στηρίζει το σχέδιο έκθεσης που προετοίμασα. Αυτά για την κυρία Κρέλ. Αν θέλετε όμως να λάβετε το λόγο εσείς, ε, με τα χαράς. Κυρία Ράιντκε, είστε σκιώδης συγγήτρια. Ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να please use your headphones because I I plan to, to speak in my mother language in Greek. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ διπλά και για την εισήγησή σας με την οποία είμαι σύμφωνος. Ε, συμφωνώ με την πρόταση που μας κάνατε να εγκρίνουμε χωρίς τροποποιήσεις την πρόταση που μας κατέθεσε η Κομισιόν. Ε, έχουμε ήδη τα, μια εμπειρία από το πώς λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός στο ΠΑΠ το προηγούμενο χρονικό διάστημα χωρίς να προσθέσει επιβάρυνση στον κοινοτικό προϋπολογισμό με μια πρόταση δημοσιονομικά ουδέτερη έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να τα πάει καλύτερα στον τομέα των επενδύσεων αλλά και δημοσιονομικά και στον τομέα της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων από ό,τι προέβλεπε η Κομισιόν, το Συμβούλιο και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Άρα από τη στιγμή που έχουμε μια εμπειρία ότι αυτό το πράγμα δουλεύει θετικά και από τη στιγμή που αυτό δεν επιβαρύνει τους Ευρωπαίους φορολογουμένους καθώς είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και αφορά στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα και σήμερα είναι μόνο η Ελλάδα νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάθε λόγο να στηρίξει την ε, πρότασή σας ε, η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις εφόσον εφαρμοστεί. Κατά συνέπεια και προσωπικά αλλά και η πολιτική μου ομάδα στηρίζει την ε, πρόταση τη δική σας κυρία Μιχαήλοβα και ζητά να εγκρίνουμε την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε και από πλευρά μας πρέπει να πω ότι υποστηρίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας και Προέδρου της Επιτροπής ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για χώρες ε, που έχουν ε, κρίση οικονομική και χρηματοπιστωτική να ε, μπορούν να αξιοποιούν τα κονδύλια αυτά ως τελευταία καταφυγή για επενδύσεις. Το είδαμε στην Ελλάδα και την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική σας εισήγηση είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνο και το υποστηρίζουμε. Ωστόσο, πιστεύω ότι κάτι θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτό είναι ε, ο συντελεστής συγχρηματοδότηση που έχουμε στην πολιτική συνοχή, ε, μακροπρόθεσμα, έχει κάποιο νόημα και θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πώς γίνεται κτήμα αυτό το ζήτημα των κρατών μελών και των περιφερειών. Αν δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση, εντάξει, συμφωνούμε, αλλά να μην γίνει αυτό τώρα κοινή πρακτική και ε, μέθοδος ε, ενίσχυσης ε, και παράκαμψη τη χρηματοδότηση και συνυπευθυνότητα, γιατί δεν θα το θεωρούν δικό τους πρόγραμμα οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη και μπορεί να μην αναλαμβάνουν και τις ευθύνε οι περιφερειακές αρχές στον βαθμό που θα τους αναλογούσα και κάτι τέτοιο δεν το επιθυμούμε. Και ένα τελευταίο που θέλω να αναφέρω, γιατί θα πάει προσωπία στην Ελλάδα ε, την επόμενη εβδομάδα, μπορούμε να συνδέσουμε και αυτά που θα δούμε εκεί με τις εμπειρίες εδώ της Επιτροπής, να δούμε ποιες είναι ε, οι απόψεις των τοπικών αρχών, τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και προσβλέπω πάρα πολύ σε αυτή την επίσκεψη να το συζητήσουμε με τους εταίρους μας εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο, παρακαλώ. Grazie Πρόεδρε, ευχαριστώ και σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε αναγκασμένοι να θυρίσουμε θετική την πρόταση της Επιτροπής, ακριβώς όπως έγινε και πέρσι για την προκαταβολή της ε, οικονομικής βοηθείας προς την Ελλάδα και είπαμε ε, ότι δεν μπορούμε να πούμε όχι και ε, στην χρηματοδότηση προς την Κύπρα. Οπότε θα πρέπει δημοσιονομικά να ακολουθήσουν αυτά τα οποία πρέπει και θα έχουμε την χρηματοδότηση, είπαμε, βάσει του άρθρου 120 και είπαμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί για την Κύπρο στις 30 του 2017. Τώρα όσον αφορά το άρθρο 24, όπως ξέρετε ήδη, Ρωμανία, Ελλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος και Ελλάδα ε, ε, είναι επιλέξιμες ε, γιατί κάνανε αυτά τα προγράμματα οικονομικής δημοσιονομικής προσαρμογής βρίσκεται σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα η Ελλάδα και θα βρίσκεται σε αυτή την ε, θέση, είπαμε, μέχρι το, τρίτο, ε, μέχρι, το δεύτερο εξάμεινο του 2018. Οπότε είπαμε ότι θα γίνει μέχρι τότε αυτή η χρηματοδότηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτά τα οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνάδελφοι για τις πληρωμές σύμφωνα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα είπαμε ότι έχουμε το άρθρο 23 το οποίο είναι διαβόητο και άρα υποχρεούμεθα να συμφωνήσουμε και όπως είπαν και οι πράσινοι ε, συνάδελφοι από τους πράσινους θα πάμε σύντομα στην Ελλάδα. Εκεί θα συζητήσουμε τη ρίζα των προβλημάτων και ελπίζω όταν γίνει αυτή η αποστολή να καταλάβουμε, να έχουμε μια αντίληψη των ε, πραγμάτων, να δούμε τι γίνεται με τις δημόσιες επενδύσεις και με την ε, πολιτική λιτότητα. Να δούμε τις τροπολογίες και Ευχαριστούμε για το έργο σας, Πρόεδρε. Ο κύριος Φανίστερα. εξ ονόματος του κυρίου Αρήμαντ που είναι ο δικός μας σκιώδης, μιλώ, έπρεπε να φύγει γιατί τον κάλεσε ο βασιλέας του Βελγίου. Οπότε σκληρή επιλογή και δίλημα. Αυτά είναι διλήμματα. Αλλά ε, δεν διαφωνεί με την πρότασή σας. Ε, το θέμα πάντα είναι το timing, έτσι, το χρονοδιάγραμμα. Μας είπατε ότι θα κάνουν γνωμοδοτήσεις άλλες επιτροπές και πολλές. Έκον λέει, δεν θυμάμαι ποιες άλλες. Αλλά τελικά, η τελική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί. Δεν μπορούμε καν να διαβάσουμε τις νομοδοτήσεις τους ακόμα. Και εμείς ε, βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν είναι πάρα πολύ διαφανή όλα αυτά που κάνουμε εδώ, έτσι δεν είναι. Ξέρω εγώ θέλω να έχω λίγο περιθώριο να διαβάσω τουλάχιστον τι νομοδοτήσει των άλλων επιτροπών και μετά να αποφασίσω. Δεν διαφωνώ. Καθόλου. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Απλώς, ξέρω εγώ. Αν ήμουν εγώ συντάκτη νομοδότης σε άλλη επιτροπή και λάμβανε ε, η επιτροπή απόφαση ερήμην μου και χωρίς τροπολογίες, πώς θα το έπαιρνα. Δεν ξέρω, μπορεί να συνοφριωνόμουν, κάπως να δυσανασχετούσα. Αφήστε δε που είναι και πάρα πολύ βιενικό αυτό. Thank you very much. Uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσέλα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι μέλος όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και δεν μπορώ τόσο εύκολα να αλλάζω ε, που κάμισο όταν αλλάζω επιτροπή και ιδιότητα. Και θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό οι ελόγω χώρες έχουν αξιοποιήσει αυτές τις διευκολύνσεις και τις εύνης που έχουν, γιατί είναι χρόνια τώρα και πώς το χρησιμοποίησαν. Βέβαια η Ελλάδα είναι έκτακτη περίπτωση και την βάζω έτσι λίγο στην άκρη. Είναι ακόμα στο μηχανισμό στήριξης και σταθερότητας. Η κατάσταση είναι όλους διάσωσα που έχει να αντιμετωπίσει. Οπότε είναι δικαιολογημένο από ό,τι φαίνεται να βοηθήσουμε τη χώρα και να τη διευκολύνουμε λίγο και για το μέλλον. Βέβαια, η κατάσταση αλλάζει για την Κύπρο. Ε, βγήκε από το πρόγραμμα στήριξη και μάλιστα βιαζόταν πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση οικονομική δεν είναι και τόσο χάλια. Και τώρα όταν μιλάμε για πάνω από 90% ε, του ΑΕΠ, ε, κατά μέσο όρο, είναι εντάξει. Κάτι που μου κάνει εντύπωση στην Κύπρο και που με ενοχλεί είναι ότι μόλις βγήκε από το πρόγραμμα στήριξης άλλαξε το φορολογικό τη σύστημα. Και ε, πέρυσι έδωσε φορολογικέ ελαφρύνσεις ε, non-dom program, resident but not domiciled, για κάποιους που δεν ζουν στην Κύπρο, που έχουν έδρα, που δεν είναι καν ε, πολίτες της Κύπρου, έχουν έδρα, ξέρω, ένα διαμέρισμα ιδρύουν εταιρεία με δύο κλικ ε, στο ποντίκι, αυτό γίνεται αμέσω και για 17 χρόνια έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις και μάλιστα φορολόγητο και ατέλεια για τα κέρδη που μεταφέρουν εκεί. Χρησιμοποιείται αυτό ε, για φοροαποφυγή εις βάρος του Ευρωπαίου πολίτη και όπως λένε οι ειδικοί, είναι καλύτερο το πρόγραμμα που προτείνει η Κύπρος από αυτό που προτείνει η Μάλτα στους επενδυτές. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Μήπως είναι λίγο άδικο, μήπως είναι λίγο στρέβλωση του ανταγωνισμού αυτό απέναντι σε άλλες χώρες. Όταν θες να προσελκύσεις έτσι ε, έσοδα ε, για λόγους φορολογικούς από κέρδη που έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Δεν μου φαίνεται ότι πάει τόσο χαλιά λοιπόν. Σε ό,τι αφορά επίσης τις δαπάνες στην Κύπρο, στην τελευταία προγραμματική περίοδο, δεν χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη διαφάνεια το νησί, στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα κονδύλια αυτή τη στιγμή στάνουν στην Κύπρο. Μου λείπει λοιπόν πληροφόρηση που δεν έχω αυτό τον καιρό και αυτά που έμαθα δεν με χαροποιούν πάρα πολύ, ούτε με κάνουν να τείνουν να εγκρίνω τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συγχρηματοδότηση στην Κύπρο. Όποιο παίρνει λεφτά από άλλους με υπομορφή φόρων και έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, από ό,τι φαίνεται δεν έχει και καμιά τρομερή ανάγκη στον προπολογισμό και δεν χρειάζεται διευκόλυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσεν, έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρότασή μου είναι ίδια με την πρόταση της εισηγήτριας, γι' αυτό τη, στηρίζω ως και όδης εισηγητής. Δεν ξέρω τις ακριβείς λεπτομέρειες της πρότασης, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι καμιά φορά η συγχρηματοδότηση δεν ε, πρέπει να προσμετράται μόνο με χρήμα. Πολλές φορές έχει να κάνει με στρατηγικές επενδύσεις και οι στρατηγικές επενδύσεις ενδεχομένως είναι και κοινωνικές επενδύσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιφερειακά ταμεία, κοινωνικά ταμεία. Η στήριξη μπορεί να έχει εθελοντική μορφή. Πώς λοιπόν μπορείς να ποσοτικοποιήσεις, να μετρήσεις την εθελοντική εργασία, όταν κινητοποιούνται οι πολίτες ή οι κάτοικοι ενό χωριού ας πούμε. Πώς μπορείς να το θεωρήσεις αυτό συγχρηματοδότηση. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγουμε, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Δεν έχουμε λεφτά, αλλά μπορούμε να δώσουμε την εργασία μας. Εθελοντικά. Και πιστεύω πως πολλές φορές αυτό είναι πιο σημαντικό από το χρήμα και θα πρέπει να θεωρείται συγχρηματοδότηση αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ε, θέση του Συμβουλίου. Έχουμε έναν εκπρόσωπο της Προεδρίας της Σλοβακίας και θα δώσω αμέσως το λόγο για να μας πείτε τη θέση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ενβέντοβα ονομάζομαι, εκπροσωπώ την ε, Σλοβακική Προεδρία. Εκ μέρου του Συμβουλίου θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου, την πρότασή σα να προχωρήσουμε εγκρίνοντα την πρόταση τη Επιτροπή. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου προ το παρόν. Αναμένουμε την έγκρισή του στο, ε, μέσα στο μήνα και αναμένουμε επίση η απόφαση να εγκριθεί χωρί τροποποίηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπέρκοβιτ, ο οποίο θα μα ε, παρουσιάσει την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, η οποία πιστεύω πως αντικατοπτρίζει πολύ πιστά την θέση της Επιτροπής. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο από τα συμπεράσματά σας. Το πρώτο είναι ε, τα εστιασμένα μέτρα που αναφέρετε και εσείς στην έκθεση. Δεν αφορούν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά ε, επιλέχθηκαν για τα κράτη-μέλη αυτά, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικά συνθήκες ε, και αναφέρομαι στο top-up ε, σε ό,τι αφορά την Κύπρο και εν είδη απάντηση στον κύριο Τσέλερ, θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση στην Κύπρο οικονομικά το 2014 και το 2015 ήταν πάρα πολύ κακή. Γι' αυτό και ε, έγινε η πρόταση της Επιτροπής. Μαζί με την Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος μέλος όπου η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις μειώνονταν. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει πολύ καλός λόγος να επεκταθεί ως τελεστή συγχρηματοδότηση και ε, επίσης τα άλλα θέματα που θα ασχοληθούμε στο μέλλον. Τώρα, όπως αναφέρατε στην έκθεσή σας, οι προτάσεις αυτές δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό. Έχει να κάνει με front-loading πληρωμών, έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε την ρευστότητα σε καιρούς δυσκολίας. Αυτά ως προς το top-up. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια που άκουσα. Να πω καταρχάς ότι συμφωνώ απόλυτα με το ότι η συγχρηματοδότηση είναι στον πυρήνα της πολιτικής συνοχής. Είναι ευθύνη των κρατών μελών και των περιφερειών της τοπικής περιφερειακής αυτοδιοίκησης σίγουρα, δίχως άλλο. Και όταν θα επισκεφτούμε την Ελλάδα σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ακριβώς ε, γίνεται, πώς ακριβώς δουλεύει το πρόγραμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε αυτό, δεν αμφισβητούμε ε, το μοντέλο της συγχρηματοδότησης καθ' αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, όπως την αντιλαμβάνομαι, μία πρόταση που στηρίζει τη διαδικασία της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και αυτό είναι η απάντησή μου στον κύριο Τσέλερ. Έχετε δίκιο, μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το φορολογικό θέμα στην Κύπρο. Η πρότασή μου όμως αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Δεν αφορά την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο γενικότερα. Στηρίζουμε την διαδικασία και την υλοποίηση της πολιτικής ε, συνοχής και των έργων σχετικών με αυτή στην Κύπρο και την Ελλάδα. Στηρίζουμε την προσπάθεια για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε αυτές τις χώρες. Και αυτός είναι ο λόγος για την γνωμοδότηση, αυτός είναι ο λόγος που το συζητάμε σήμερα και αυτός είναι ο λόγος που προτείνω να μην τροποποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα κάνουν οι άλλες επιτροπές. Εμείς όμως είμαστε υπευθύνοι για τη δική μας γνωμοδότηση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό μόνο. Και πιστεύω πως είναι λογικότατο. Έχει γίνει ήδη στο παρελθόν μια φορά για την Ελλάδα και μπορούμε, επειδή είδαμε πολύ θετικά αποτελέσματα, να συνεχίσουμε. Εάν υπάρξουν προβλήματα θα έχουμε τη δυνατότητα να το διερευνήσουμε, να ρωτήσουμε τις ε, τοπικές αρχές, τους αρμόδιους φορείς στη χώρα, στην Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση όμως, το σύνολό της, πιστεύω πως είναι αρκετά εξισορροπημένη. Θεωρώ, συγγήτρια. Γι' αυτό λοιπόν η στάση που προτείνω είναι να μην τροποποιήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Συμφωνούμε λοιπόν να μην τροποποιήσουμε την πρόταση ή υπάρχει επιθυμία να γίνουν τροποποιήσεις, να υποβληθούν τροπολογίες. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βανίστα Θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Δεν έχουμε ακόμα... Ε, ε, εμείς δεν κάνουμε γνωμοδότηση εδώ, κάνουμε την έκθεση, έτσι. Είμαστε επί της ουσίας. Τι γίνεται με εκείνους που γνωμοδοτούν. Δεν θέλουμε να δούμε το περιεχόμενο της νομοδότησης άλλων επιτροπών πριν ψηφίσουμε. Εντάξει, να, να ψηφίσουμε ότι δεν θα κάνουμε τροπολογίες, αλλά προσοχή να περιμένουμε τις νομοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπα προηγουμένως. Συμφωνώ καταρχήν, αλλά με τη διαδικασία έχω πρόβλημα. Okay. Οι γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών θα επισυναυθούν στην έκθεση και δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε τροπολογίες και ε, θα τα ξαναπούμε και θα επισυνάψουμε όλες τις νομοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών και θα λάβετε γνώση αυτών. Θα ενημερωθείτε. Εντάξει, είμαστε. Επίσημα θα ψηφίσουμε την άλλη φορά στην επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Προχωρούμε. Next, uh, Επόμενο θέμα. Έκθεση της πρωτοβουλίας του κ. Πανίστερόη. Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Όχι, δεν είναι ιδέας πρωτοβουλίας. Ζητάει συγγνώμη, Πρόεδρε επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του ο εισηγητής, βελτιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαθετικών και Επενδυτικών Ταμείων, αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16, παράγραφος 3. των κοινών ε, κανονιστικών διατάξεων. Στις 13 Ιουλίου είχαμε ανταλλαγή απόψεων και ο κύριος Βανίστε Ρόι μοιράστηκε τις ιδέες του μαζί μας και ε, το κύριο συμπέρασμα των επαφών που είχε με τους ενδιαφερόμενους ε, για τα επιχειρησιακά προγράμματα όπως ε, ζητεί το άρθρο 16 παράγραφος 3. Στην τελευταία συνεδρίαση και στην ακρόαση της 15ης Ιουνίου ο εισηγητής εστίασε σε κάποια βασικά σημεία από τα οποία μπορούμε να λύσουμε διδάγματα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Σήμερα ο κύριος Μανίστερο θα μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής του. Προτείνω ε, προθεσμή για την κατάθεση τροπολογιών την 5η 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά μπορώ να σας πω ότι με βλέπουν και οι ε, δικοί μου, γι' αυτό μιλάω Ολλανδικά και με ακούνε ε, στην εκλογική μου περιφέρεια. Ε, όπως είπε και η Πρόεδρος, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων, είχαμε μια ακρόαση, ακούσαμε διάφορα και τα έχουμε σημειώσει. Ξέρω ότι διάφορες πολιτικές ομάδες εδώ στην Επιτροπή έχουν και ίδιες δράσεις και δραστηριότητες για να αντιδράσουν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη έκθεση που μπορείτε να διαβάσετε τι έγινε στην περίοδο 2014 με 2020, τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια μαζί με τα τοπικά, περιφερειακά, κρατικά και καμιά φορά και ιδιωτικά, ακόμα και των οικοκυριών χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, για ε, θέσεις εργασίας και τα λοιπά και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα καλό λοιπόν χρονικό σημείο και μια ωραία στιγμή για να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και να τα αξιολογήσουμε που είναι στο κάτω-κάτω και δική μας δουλειά στην Επιτροπή μας για να φτάσουμε ε, στην Ολομέλεια και να ληφθεί απόφαση. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις. ένα έγγραφο εργασία. Ε, υπάρχει που σημειώνει κάποια πράγματα τα οποία έχω συμπεριλάβει και εγώ στην πρώτη μου πρόταση και πολύ μου χρησιμεύσαν. Ε, πέρα από αυτό όμως θέλω να πω μερικά πράγματα. Πρώτον, έχουμε τα διάφορα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία ως μέσα, ως εργαλεία που είναι χρήματα των φορολογουμένων και χρησιμοποιούνται όχι μέσα σε ένα εργαλείο, αλλά διαχέονται σε όλα τα κράτη-μέλη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ε, συμμετοχή περιφερειών και πόλεων. Είναι πραγματικά ευρωπαϊκά αυτά τα μέσα και τα εργαλεία. Δεν είναι κάτι για ένα συγκεκριμένο κλάδο, αλλά είναι εγκάρσια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ζήσαμε κρίσεις. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είχαν εξαντλήσει το περιθώριο που είχαν για τις δημόσιες δαπάνες από τον κρατικό προπολογισμό, τον τοπικό ή τον περιφερειακό και η μόνη λύση ήταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και λόγω των κρίσεων και λόγω των δημοσιονομικών ε, ε, συμφωνιών που είχαν λόγω των ελλημάτων. Ήταν δεσμευμένε οι χώρε αυτέ και δεν μπορούσαν να επενδύσουν, αλλά ήταν σε πάρα πολύ δεινή θέση. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν στην έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ πήγε αυτό το εγχείρημα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο το εργαλείο και πολύτιμο. Το δεύτερο που μπορείτε να δείτε είναι πού πηγαίνουν τα λεφτά. Είπαμε και ε, στους ε, ε, κανονισμούς ότι δεν το μοιράζουν τα κράτη-μέλη κατά το δοκούν ανάλογα με το αγαπημένο τους θέμα, αλλά υπάρχουν και προτεραιότητες. Θα πρέπει η γνώση να μεταφέρεται σε θέσεις εργασίας, σε εκπαίδευση, σε κατάρτιση κτλ. Η γνώση και η καινοτομία. Αλλά αυτό θα πρέπει να ενισχύει το κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα ή γενικότερα το επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτά είναι τα δύο πρώτα. Ε, και κλασική επιλογή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να πει ότι ε, η τεχνολογία της πληροφορικής είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ όλοι έχουμε ένα iPhone και επικοινωνούμε, αλλά ε, μεταφέρεται σε όλους τους τομείς. Κοιτάξτε τι κάνουμε, τα τραπεζικά μας, τα διάφορα ε, θέματα υγείας, ε, διεκπαιρεώνουμε εκπαίδευση, παιδεία, παντού υπάρχει πληροφορική, μέχρι και στην ιατρική και στα συστήματα υγείας τα στοιχεία των ασθενών. Μετά, ό,τι έχει να κάνει με την αηφορία στο περιβάλλον και το βιώσιμο περιβάλλον. Ενέργεια, ενεργειακή μετάβαση δηλαδή, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όλα αυτά τα θέματα, ε, καλύτερη στέγαση και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα ρυθμίζει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επίσης μια σειρά στόχων έχει να κάνει με ε, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν θα πρέπει κανείς να αφήνεται στην άκρη στο περιθώριο της κοινωνίας. Ε, και θα πρέπει αυτά να λαμβάνονται ως αποφάσεις πολύ κοντά στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να τους δίνεται μια προοπτική που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτούς τους καιρούς. Και κάτι άλλο που είναι η περιφερειακή διάσταση, η εδαφική διάσταση, η διασυνοριακή, που ε, θα πρέπει να μαθαίνουμε καλύτερα και πιο γρήγορα ένας από τον άλλον και να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και ε, το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ θετικό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται, ξέρω εγώ, άνωθεν από τις Βρυξέλλε, που είναι κάτι το απόμακρο και σκοτεινό, αλλά είναι στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική κοινωνία και κοντά στου ανθρώπους. Αυτά ήθελα να σας πω. Να μην χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας στην Ευρώπη, να διατηρήσουμε ψηλά όλα αυτά τα εργαλεία. Επόμενο σημείο. Βλέπετε ότι η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παρούσα το συζητάμε. Ε, είχαμε πάει με διαφόρους και από όλες πολιτικές ομάδες την τελευταία τερκουάς εβδομάδα στη Silicon Valley. Εκεί να δείτε πώς οριάζει η τεχνολογία, ε, τι εξελίξεις έχουμε, οι χώρες της Ασίας, ε, τι κάνουν με το λογισμικό, με τα μαθηματικά, με τους νέους, πώς εκπαιδεύουν ε, πώς τους καταρτίζουν, τι δυνατότητες υπάρχουν για την οικονομία, για τους κοινωνικούς στόχους, για τις υπηρεσίες. Είναι πράγματα θαυμαστά. Και θα πρέπει να προσέξουμε στην Ευρώπη να μεταφέρεται αυτή η γνώση και να δημιουργεί θέσεις εργασίας και σε θέματα τεχνολογίας πληροφορίας. Το ταμείο αυτό λοιπόν, ή τα ταμεία καλύτερα που είναι πέντε, ε, είναι στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας Έχουμε 10 συμφωνίες ε, για να αποδώσουμε, ή 11 δεν θυμάμαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και ε, εργασίας. Δεν είναι τίποτα καινούριο, τίποτα διαφορετικό, αλλά θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους αυτά. Ας πούμε, ε, παράδειγμα το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το συζητήσαμε το πρωί. Τα επενδυτικά ταμεία ή ορίζον 2020 όταν πρόκειται για την αριστεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, είναι ε, ξεχωριστά εργαλεία τα οποία όμως τέμνονται ή εφάπτονται. Και τη συζήτηση αυτή την κάναμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτέλους καταλαβαίνουν καλύτερα και περισσότερο αυτά τα πράγματα από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Γιατί, διότι έχουμε από κοινού τώρα προβλήματα με τον Brexit και τους μπελάδες που μας έχουν βρει στα θέματα της ασφάλειας και έχει απόλυτη σημασία ε, ο Ευρωπαίος πολίτης να ζει την αλληλεγγύη στο πετσί του. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργεί ε, συνδέσεις ε, και αλληλεγγύη. Και πιάνουν τόπο αυτά τα ταμεία, αν το συγκρίνουμε με λίγα χρόνια πριν, έχουμε και μια νέα ευκαιρία επιτέλους να το συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε καλύτερα. Έχω και επικριτικά και αρνητικά μόνο σιγά μη δεν είχα. Η περίοδος αυτή ε, άργησε να ξεκινήσει. Τα λεφτά υπήρχαν, αλλά για να πάρει μπρος αυτή η ιστορία χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και χάσαμε καιρό. Και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, θα γίνουν και κάποιες τροπολογίες. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν αυτό και θέλουμε να τα προσαρμόσουμε για το μέλλον, να αρχίζουμε νωρίτερα μαζί με το Συμβούλιο για να επιταχύνεται η έναρξη αυτή η κίνηση και στο νέο κανονισμό και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος όπου τραβάει σε μάκρος αυτή η ιστορία με ατέρμονες συζητήσεις και πάει λέγοντας. Αλλά γρήγορα να βάζουμε το χέρι στην ε, Το δεύτερο πρόβλημα είναι η περιπλοκότητα. Είναι περίπλοκα. Από τη μια έρχεται η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εμεί οι ίδιοι και θέλουμε performance based, λέει, ε, με βάση τις επιδόσεις να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, όχι να δίνουμε λεφτά σε φακέλους και τους λέμε κάντε τίποτα καλά πράγματα εκεί πέρα. Όχι, βάσει των επιδόσεων και θα πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις και αποτέλεσμα. Ε, και για να είναι αμοιβαία επωφελέ αυτό. Ρωτήσαμε και τους αρμόδιους στη Γενική Διεύθυνση Ραγκιό. Χρειάζεται μία εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Αυτό χρειάζεται χρόνο για να ελεγχθεί. Αλλά ευτυχώ αυτό τον καιρό προχωρούν σε μια απλοποίηση του συστήματος και τα λέει και η έκθεσή μου. Τρίτο σημείο έτσι κριτικής και τελευταίο στην εισαγωγή είναι ότι η έλλειψη προβολής Υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε ένα κόμπο εκεί πέρα. Όχι ένα κόμπο στο λαιμό, αλλά ένα κόμπο στην επικοινωνία. Έχουμε ένα προπολογισμό και απ' την άλλη τώρα που ε, σηκώνουν κεφάλι οι εθνικισμοί και οι λαϊκισμοί σε πάρα πολλές χώρες, θα πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Στον Ρωμαίο Βασίλειο, βλέπετε τι γίνεται. Στην Ουαλία που έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από εμάς ψηφίσανε Brexit θέλουν να φύγουν. Γιατί λέει δεν μας βοηθάει η Ευρώπη καθόλου. Αυτά είναι διαστρέβλωση, ο κόσμος δεν τα ξέρει και φταίμε και εμείς. Κάτι κάναμε στραβά στην επικοινωνία. πέρασαν και παρήλθαν οι εποχές των ε, παχιών Ελλάδων που ε, ανέβαινε ε, ο προπολογισμό και η ευημερία και όλοι είχαν περισσότερα λεφτά. Τώρα που έχουμε τους εθνικισμούς, όλα αυτά τα προβλήματα, το Brexit, χρειάζεται διαφορετική επικοινωνία. Και από εκεί ξεκινάω. Που λέω, μα τι στο καλό, κάπως αλλιώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και αυτό μέσα στα project, μέσα στα έργα και τα κοινωνικά έργα και να ξέρει ο καθένας ότι α, βρήκα δουλειά επειδή υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα ε, πρόγραμμα και χαίρομαι και μπράβο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν τα λέμε, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να βρίζουμε τα διάφορα έργα ότι είναι πολύ γραφειοκρατικά και πρέπει να σταματήσουν, αλλά στην επικοινωνία χωλένουμε. Και τελευταίο. Είμαι πρόεδρος στην ε, εξεταστική επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον σε μια ε, επιτροπή ενό διαγωνισμού ε, για τις ευρωπαϊκές πόλεις για το πώς διακρίνονται και δίνουμε διάφορα αστέρια εκεί πέρα τους χειροκροτούμε όταν έρχονται και τους τα απονέμουμε αλλά όλα αυτά πρέπει να προβάλλονται Καλό είναι να λέμε πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνονται καλύτερα διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να τα προβάλλουμε όλα αυτά ε, και ε, μαζί με τα κράτη-μέλη και πώς εκτελούνται αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει λίγο να τα γυαλίσουμε, να λάμπουν περισσότερο, να, να ακτινοβολούν. Κάποιο είπε ότι είμαστε πράσινη πόλη τη Ευρώπη. Ε, διότι όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει την αποκομιδή και την επεξεργασία των αποβλήτων. Το ξέρει αυτό που έχει γίνει πράσινη πόλη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω σε όποιον βλέπω. Αλλά δεν το ξέρει κανεί. Βάζει κάποιο μια σφραγίδα που είναι η σημαία με τα στεράκια και χαιρετίσματα και μετά από τρία χρόνια πρέπει να έρθει να το ξύσει γιατί έχει σκουριάσει. Πρέπει να βγάλει το πράσινο για να φανεί το μπλε από κάτω και τα αστεράκια και έχει πεταχθεί η Ευρώπη στο κάλαθο των αχρήστων. Το 10% των προγραμμάτων πηγαίνει στην προβολή. Δηλαδή, be good and tell it. Να, να είσαι καλό να το λε κιόλα, να το μαθαίνει ο κόσμο, να το διαφημίζει. Αυτά. Την άλλη εβδομάδα για να τελειώσω θα πάμε μαζί με την πρόεδρο σε μια διάσκεψη της Σλοβακικής Προεδρίας για το μέλλον της συνοχής και εκεί θα τα πω και αυτά. Να δούμε πώς θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο να φτάνουμε στον πολίτη τα κακό κείμενα, εντάξει δεν χρειάζεται να τα τονίζουμε, αλλά να λέμε και τα καλά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ λοιπόν οι δικές σας απόψεις, η δική σας συνεισφορά Και ε, θα ξαναπούμε τον Οκτώβριο. Έχουμε δύο συνεδριάσεις στο Στρασβούργο ε, με τους Κιώδης. Κάποια στιγμή θα βρούμε χρόνο. Και για αλλαγή ε, και καταξαίρεση τα είπα και Ολλανδικά σήμερα, Πρόεδρε. Thank you. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για το συνεχισμό τους Κιώδης ηγητές. Κυρία Βέστολ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, όντως Τώρα είμαι η συγκήτρια κανονική και άριστα προετοιμασμένη. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης μάλλον του Λάμπερτ Μο ε, Νίστελροι με χαροποιεί γιατί η Προεδρία του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή συνεργάζεται μαζί μας καλά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι αυτή η καλή συνεργασία. Ε, έχω κάποιες παρατηρήσεις για το σχέδιο έκθεσης που δεν αντιτίθενται σε αυτά που θα πω στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα να πω αυτής εξ αρχής ότι δεν μου είναι ακριβώς αφήσει η στόχη ή ο στόχος αυτής της έκθεσης. Εάν δηλαδή με αυτήν την έκθεση θέλουμε να αξιολογήσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δω τον τίτλο τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Ή εάν θέλουμε να ε, προετοιμάσουμε το έδαφος για το τι θα γίνει μετά το 2020. Την προηγούμενη φορά νομίζω το είπα κιόλα ότι δεν θεωρώ αντίφαση ακριβώς μετά από την ε, έκθεση του κ. Βανίστελ να μιλήσω έτσι. Νομίζω πως η έκθεσή του είναι πάρα πολύ καλή τα κατάφερε και να μας κάνει μια ανασκόπηση, αλλά ταυτόχρονα να κοιτάζει και προς τα εμπρός. Όμως πολλές φορές αυτό οδηγεί σε συγχύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ορισμός, το, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το new period, η νέα περίοδος είναι μια αλλαγή προοπτικής, ε, αναφέρεται στην ε, τρέχουσα περίοδο στήριξης ή την επόμενη, όπως λέει στο σημείο 23. Μου φαίνονται κάπως μπερδεμένα και δεν νομίζω ότι είναι η γερμανική μετάφραση, γιατί είδα και το αγγλικό κείμενο. Γι' αυτό δεν σας κάνω την έξυπνη. Νομίζω πως ο Λάμπερτ ε, αναφέρει πολλά σημαντικά θέματα. Η έκθεση, για παράδειγμα, αρχίζει με την ορατότητα της πολιτικής συνοχής και εδώ με βρίσκει 1000% σύμφωνη, όχι 100% μόνο. Οφείλουμε πράγματι να πουλήσουμε στους πολίτες καλύτερα την πολιτική συνοχής, διότι ακριβώς αυτή η πολιτική συνοχής είναι η, επενδύση, η επένδυση του μέλλοντος και αυτό δεν το λέω πρώτη φορά, ούτε θα είναι η τελευταία. Πώς λοιπόν θα πουλήσουμε αυτή την πολιτική συνοχή, πώς θα σταθούμε ε, ενώπιον των πολιτών. Πέρα από την έκθεση, θεωρώ ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές, οι επιτροπές, όλοι όσοι εργάζονται εδώ ε, χρειάζονται να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Χρειάζεται να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, να περάσουμε στο περιφερειακό, στο τοπικό. Ε, στη Γερμανία έχουμε και άλλο επίπεδο, έχουμε και το μοσπονδιακό επίπεδο. Πρέπει να ε, κινητοποιηθούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση, έτσι ώστε να μάθουν οι πολίτες τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού, τι γίνεται όταν κάποιο βρίσκει μια δουλειά. Ποιο χρηματοδοτεί αυτήν τη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς, ε, μέσω της ε, ε, διασφάλισης ότι πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μετά, παράδειγμα, στην Πολωνία παντού. Αν πάτε θα δείτε ε, ότι υπάρχουν πινακίδες που λέει συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το, το έργο, το τάδε, το δίνα, έχει γίνει με κονδύλια κοινοτικά. Παντού στη χώρα τα βλέπεις αυτά. Και όπως είπατε κι εσείς, καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει κάνει η Ευρώπη. Όταν βλέπεις τεράστιες πινακίδες που πάνω τους αναγράφονται ποσά, αναγράφονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια για τα έργα, συνειδητοποιείς τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, ε, η θεματική συγκέντρωση, που είναι κάτι που ακούσαμε πιο πριν, είναι σημαντικό. Και στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο μάλιστα το παλέψαμε ώστε αυτή η θεματική συγκέντρωση να έχει αποτέλεσμα και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στην σωστή επένδυση των χρημάτων, δηλαδή να στηρίξουμε τις επενδύσεις, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να στηρίξουμε τους ε, σχετικούς τομείς, ε, να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή, Λάμπερτ, το είπες και αυτό εξάλλου, και πιστεύω πως σε αυτό το θέμα πάμε καλά, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως όλα είναι μια χαρά σε αυτόν τον τομέα, έτσι όπως τα διαβάζω. Μετά, βλέπω πως αυτή η απλούστευση είναι πάρα πολύ θετική, πολύ επίπεδη διακυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένας εδώ ή οπουδήποτε αλλού ότι η απλούστευση είναι κακό πράγμα. Επίσης, στο σημείο 32 αναφέρονται οι αρχές των εταιρικών σχέσεων και αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ σημαντικό. Πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή ε, εδώ και να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι καταφέραμε ένα, να, περάσουμε σε ένα σημείο, να περάσουμε μάλλον ένα ορόσημο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα πώς θα συμπεριληφθούν και άλλοι στην, στην χρηματοδότηση, πώς θα ενημερωθούν γι' αυτό στη συνέχεια οι πολίτες. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο μου αφήνει κάποιες ε, αμφιβολίες. Η σύνδεση δηλαδή με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω και τόσο. Ο ρόλος ε, δηλαδή αξιολόγηση επιδόσεων, αυτό δεν θα σε εκπλήξει η Λάμπερτ ότι με βρίσκει κάπως ε, αντίθετη. Έχω κάποιες ε, αμφιβολίες, κάποιους δισταγμούς και είναι το μόνο πράγμα που με πονοκεφαλιάζει λιγάκι στην όλη έκθεση. Μετά, πέραν αυτών, θέλω να πω ότι έχεις κάνει μια εξαιρετική έκθεση και χάρηκα πάρα πολύ που δούλεψα και που θα συνεχίσω να δουλεύω μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος και τώρα συνεχίζουμε. Και όλοι ηγητές, ο κ. Γιάκοψης. Θέλετε τον ε, λόγο για λογισμό κ. Μίλτεμπερ. Ναι, δυστυχώς και ο συνδεσμού δεν μπόρεσε να παραστεί, διότι βοηθά στο Γιβραλτάρ στον κόσμο. Οπότε να προσπαθήσω αντί γι' αυτόν να σας πω τι πρεσβεύει όσον αφορά την ε, εκθέση Λάμπερτς. Πιστεύω ότι θα, θα, θα δείτε ότι ένα σημείο στο μέλλον. Αλλά και ο Μίλτενμπεργκ εξοπλίσετε, γιατί δεν αναφέρεται η σχέση μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ε, πολιτικής συνοχής. Έτσι θα τονωθούν οι επενδύσεις. Θεωρεί. Επίσης, λέει για περισσότερη ευελιξία που θα πρέπει να δίνουν του θεματικού και τα ταμεία ήδη έχουν ε, πάρα πολλού στόχου και ευελιξία. Θα πρέπει να καλύψει κάποια ζητήματα τα οποία αναδύονται μόνο μετά την έγκριση κάποιων λειτουργικών προγραμμάτων. Επίση, ε, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία για κάποιε συστάσει που αφορούν συγκεκριμένε χώρε. Και έχουμε αυτού τους κανόνες για κρατικέ ενισχύσει μεταξύ προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών Ταμείων και ο και επίση θέλει να υπάρξει κάποια εξέταση της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έρθουν ό,τι να υπάρχουν. Επίσης λέω ότι το ΑΕΠ δεν θα πρέπει να είναι το μόνο θεμητό κριτήριο για την κατανομή των πόρων. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα κριτήρια. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Οπότε και με τον κύριο Ματές θα γίνει συζήτηση γιατί αυτή τόσο αξιόλογη έκθεση που είναι πάρα πολύ καλά στοχευμένη αλλά ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί με τις προτάσεις μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντοματό, έχετε το λόγο. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για το σχέδιο της εκθέσεως για αυτή την επίκαιρη έκθεση κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου. Πρόκειται και κάποια έκδοση όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτών των ε, διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του, του για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει 31 του 2015. Η πολιτική τη συνοχή θα πρέπει να το περισσότερη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Και τι εννοούμε, ότι θα πρέπει να πέσει φω στι απάτε. Γιατί η πολιτική συνοχή είναι το βασικό εργαλείο για τι επενδύσει στην Ένωση. Επομένω, θα πρέπει οι ιδέες και τα έργα να αξιοποιούνται και να προωθούνται. Η χρηματοδότηση γίνεται σε κάποια έργα χρήσιμα καταρχήν και με την συμμετοχή και συγχρηματοδότηση της Ευρώπης και με τους σχετικούς ε, δείκτες τότε θα θωρακίσουμε την πολιτική αυτή. Όμως είναι απαράδεκτες κάποιες καθυστερήσεις στα λειτουργικά προγράμματα όσον αφορά τις ε, δαπάνες, αλλά χρειάζεται επιτάχυνση ακόμα και με τα βασικά προγράμματα. Επίσης, το ελεγκτικό συνεδρίο διαπίστωσε ότι πάρα πολλά σφάλματα τα κολλάει η πολιτική ε, το, ή τις από άλλες πολιτικές, όπως ας πούμε τις κρατικές ε, τις κρατικές συμβάσεις. Θα πρέπει να γίνει συγκέντρωση του θεματολογίου και να υπάρχει αιρεσιμότητα εξάντε και επίσης να χρησιμοποιείται σαν κριτήριο και η επίδοση. Θα πρέπει επομένως να δούμε το θέμα της απλούτευσης που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ομάδα εργασίας που ασχολείται με αυτό θα πρέπει να γίνει ανάλυση από την Επιτροπή για τα μέτρα πλούτευσης που ήδη έχουν ληφθεί. Simplified cost options είναι ένα από αυτά τα ήδη ληφθέντα μέτρα. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο του εισηγητή θα τα πούμε στην συνάντηση των σκιωδών. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Θέλει άλλο το λόγο. Όχι. Οπότε θα δώσουμε τώρα το λόγο Στου εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κυρία Κάντρι Γουστάου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε γιατί διαβάσατε προσεκτικά το κείμενό μας. Θέλω να σας ε, αναφέρω τέσσερα τεινά, ούτω ώστε να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις αλλά και ενημέρωση γιατί οι εξελίξεις είναι καθημερινές στο θέμα αυτό. Βεβαίω. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα με το κείμενο του εισηγητή όσον αφορά τώρα την ανακοίνωση. Ε, Βεβαίω και όλα μπορούν να επιδέχονται βελτίωση και προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση να δούμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε και η ανακοίνωση να μην αφορά μόνο κράτη-μέλη ή κομισιόν. Όλοι θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ούτω ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας. Έχουμε μία πλατφόρμα που δημοσιοποιήθηκε ταυτόχρονα με τις εκθέσεις του άρθρου 16 και για πρώτη φορά τώρα εκ των προτέρων στην αρχή περίοδου προγραμματισμού μπορούμε να ορίσουμε πού θα καταλήξουμε συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ. Ανακράτος μέλος, αναπρόγραμμα και αναταμείο. Άρα μπορείτε να τσεκάρετε για τη χώρα σας ή για τις χώρες που θα επισκεφθείτε τι έχουμε υποσχεθεί να καταφέρουμε. Και με αυτή την πλατφόρμα μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Οπότε αυτή η πλατφόρμα Open Data ε, περιέχει το τι έχουν ε, δεσμευθεί να κάνουν τα κράτη-μέλη και λέμε τι θα πρέπει να πετύχουν και αργότερα πρόκειται να υπάρξει και ενημέρωση του τι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Και προχωράμε ανά έτος και βλέπουμε την πρόοδο από, αυτό το, από αυτή την πλατφόρμα. Φαίνονται και οι πληρωμές που έχουν εκταμιευθεί. Δεν χρειάζεται να περιμένετε 7 ετία ή δεκαετία. Άρα για να διαπιστώσετε εάν κάτι έχει επιτευχθεί με τα χρήματα των φορολογουμένων. Τώρα όσον αφορά το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. μία προειδοποίηση. Προσοχή, ακόμα είναι νωρίς για το ταμείο αυτό. Ξεκίνησε με επιταχύνση το Ταμείο αυτό, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Άρα, ας αφήσουμε να οριμάσουν οι εξελίξεις και τότε να συμπεράνουμε τι έχει γίνει. Τώρα όσον αφορά αυτό το διοικητικό άχθος, δεν περιέχει η έκθεσή μας τις σχετικές μελέτες. Πάντως σας ενημερώ ότι έχουμε μελέτες και θα σας τις παρουσιάσουμε. Μία μελέτη έγινε το 2010, άλλη το 12 εν ώψη της πρότασης 14-20 ενδελεχής αυτή η μελέτη και άλλη μία τώρα ολοκληρώνεται σε σχέση με την θέσπιση των μέτρων απλούστευσης από τα κρατη Αργότερα φέτος θα έχει ολοκληρωθεί και θα σας την παρουσιάσουμε αν θέλετε. Τέλος, όσον αφορά για την εκ των προτέρων χαιρεσιμότητα πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν κάποιες προθεσμίες για τα προγράμματα δράσης προβλέπονται σχεδόν για το τέλος της χρονιάς η Επίτροπος Κρέτσου τέλος Αυγούστου ενημέρωσε τη Γερμανία για το 25% της ερεσιμότητας που δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα έχουμε το 34% των πραγμάτων που έχουν ολοκληρωθεί. πάση περιπτώσει, μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε σχεδόν το σύνολο των όσων θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος. Κύριε Φανίσταλο, θέλετε το λόγο. Βέβαια, βέβαια. Σύντομα, σύντομα. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Τα παρακολούθησα αυτά που είπατε. Θα κάνουμε ε, τροπολογίες όλοι, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε όλοι την ίδια πορεία και χαίρομαι γι' αυτό. Ένα σημείο μόνο. Η κυρία Βέστφαλ είπε κάτι ε, για ε, το αποθεματικό επιδόσεων. Είπε ότι δεν το έχουμε τηρήσει με τον τρόπο της. Ε, και το κοινοβούλιο ολόκληρο. Γιατί δεν παίρνει μια στάση πιο ισχυρή, πιο στεναρή. Τι είναι αυτό το αποθεματικό, έχουμε δεσμευτεί για ένα ποσό για τη συνοχή και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τότε είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε ένα σύστημα όπου θα συμφωνήσουμε εκ των προτέρων ποια είναι τα αποτελέσματα. Εξάντε και εξ εκ των προτέρων και εκ των υστέρων θα έρθουμε να τα κοιτάξουμε αν τα κάναμε καλά η μεγάλη καινοτομία τώρα ποια είναι. Διατηρούμε στην άκρη κάποιους πόρους έτσι ώστε να επιβραβεύουμε μια χώρα που έχει ιδιαίτερες επιδόσεις. 6%. 21 δισεκατομμύρια ευρώ είναι στην άκρη. Το σύστημα αυτό συμφωνήθηκε έτσι ε, ώστε να γίνεται κάπου αξιολόγηση ενδιάμεση στη, μέση και μετά. Και βγαίνουν οι καλοί και επιβραβεύονται και δεσμεύονται για την περίοδο, αλλά ε, η ε, εκταμείευση θα γίνει την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μα είναι τόσο μεγάλη η φιλοδοξία που μπαίνει στα έργα αυτά. Γιατί εκείνοι που το 2018 δείχνουν ότι είναι τέλεια ε, όλα στην εκτέλεση και είναι τα υποδείγματα και που πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, και εκείνοι που δημιουργούν θέσεις εργασίας και βλέπουμε ότι ε, ε, διακρίνονται και οι πόλεις και μπορούν να τα κάνουν όλα καλά για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον κόσμο γιατί τους τα στερούμε αυτά. Γιατί δεν λέμε ότι για αυτά τα κράτη-μέλη που τα έχουν τελειώσει, γιατί δεν μπορούμε να τα εκταμιεύουμε, γιατί δεν αρχίσαν όλοι καθυστερημένα. Εκεί χρειάζεται κάποια ευελιξία. 21 δισεκατομμύρια έχουμε βάλει στην άκρη και θα το δούμε μετά το 2021. Μα τι είναι αυτό, τι χαλαρότηση είναι αυτή και τι ε, συμπεριφορά. Η κυρία Βέστφαλ ε, έχει δίκιο ότι θα πρέπει να έχουμε πιο επιθετική ε, συμπεριφορά. Να ρωτήσουμε το Συμβούλιο, πού το πάει, την Κομισιόν, τι προθέσεις έχει. Έχουμε προχρηματοδότηση, ακούσαμε για την Κύπρο κτλ., όταν έχουμε προβλήματα είμαστε πρόθυμοι να βοηθούμε. Αλλά όταν πάνε τα πράγματα καλά και έχουμε καλή προοπτική, δεν ε, δείχνουμε τον ίδιο ζήλο και την ίδια προθυμία, ούτε την ίδια ταχύτητα. Εντάξει, αυτή είναι η πρόκληση, κυρία Βέστφαλ. Να φέρουμε μια πρωτοβουλία. Κάντε έκθεση πρωτοβουλίας, υποβάλλετε κάτι. Στη δική μου έκθεση δεν γίνεται αυτό γιατί είναι το άρθρο 16 παράγραφος 3 η κατάσταση των πραγμάτων. Αλλά δεν σας εμποδίζει κανείς να κάνετε κι εσείς κάτι από πλευρά σας. Αυτά. Και ελπίζω φέτο σιγά σιγά να πάρει το δρόμο τη Ολομέλειας η έκθεση, έτσι να ολοκληρώνεται μέσα στο έτο. Ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, λέει η Πρόεδρο, στις 12 το μεσημέρι, την άλλη Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου. Um, here I conclude... Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η ε, ε, συνεδρίαση, αν δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, ωραία. Περίεργος πώς. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας θυμίζω, η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα την 3η 11 Οκτωβρίου 9 με 12.30 το πρωί και 3 με 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ τους Δερμηνείς. Οι Δερμηνείς ευχαριστώ την Πρόεδρο. Λήξεις για σήμερα. Σας ευχαριστώ.